Ταρέντ προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για τέσσερα λεπτά, παρακαλώ. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το χρήμα έχει σημασία φυσικά και ο χρόνος είναι χρήμα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό, είναι το εξής. Είναι τριγωνική η άσκηση του προϋπολογισμού, δηλαδή το οικονομικό έτος. Δεν το γνωρίζει αυτό το κοινό. Και ο εισηγητής πρέπει να ακολουθεί στριφνούς κανόνες διαδικαστικούς με άκαμπτη ερημηνία και πολύ συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, πολύ στενά χρονικά περιθώρια για να υπάρξουν επικοδομητικές συζητήσεις. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλώς περιμένει το Κοινοβούλιο να τηρήσει τις προθεσμίες και αν εγκριθεί η έκθεση αύριο μπορούμε επιτέλους να πούμε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, υπάρχουν ένα σωρό κανονισμοί, συμφωνίες κυρίων, διοργανικές συμφωνίες, εκτιμήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πράγματι, πράγματα που έχουν αποφασιστεί από τις προηγούμενες γενιές, από τους προκάτοχούς μας και επηρεάζουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Γιατί δεν μπορεί κανείς ούτε να ε, αυξήσει ούτε να μειώσει κονδύλια, ακόμα και όταν αυτό είναι, ε, φαίνεται είναι απολύτως απαραίτητο. Και αυτό ήταν ε, ένα και από τα πιο δύσκολα ε, πράγματα, ε, εμπόδια που συνάντησα κατά την κατάρτιση αυτής της έκθεσης. Ε, όμως, χάρη στο προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη Γραμματεία, στους συναδέλφους, στους συμβούλους, στους σκιώδεις εισηγητές και συντονιστές, χάρη στον πρόεδρο της Επιτροπής, μπόρεσα να συντάξω, πιστεύω, μια έκθεση που αποτελεί, που απεικονίζει τη συμφωνία μας είμαστε εδώ και είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να κάνουμε ε, εξοικονόμηση γιατί είναι δύσκολη καιρή έξω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πρέπει να διαχειριστούμε τις ανάγκες ε, λειτουργίας ε, του οίκου μας. Και όλα αυτά έχουν δώσει λαβή για πολύ έντονες αντιπαραθέσεις. Προσπαθήσαμε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις και ε, το κείμενο αποτελεί προϊόν της δημοκρατικής βούλησης της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό. Κάτι το οποίο πάντοτε με βρίσκει σύμφωνο όταν είναι προϊόν δημοκρατικών διαδικασιών η απόφαση. Και γι' αυτό σας καλώ να υπερψηφίσετε την έκθεση. Η Επιτροπή για τον προϋπολογισμό συζήτησε το ένα θέμα και το Προεδρείο επίσης για την εσωτερήκευση της μεταφοράς των Ευρωβουλευτών δεν έχει ε, ληφθεί η απόφαση, θα επανέλθουμε και θα αποφασίσουμε κατά πόσο θα απελευθερώσουμε τα κονδύλια ή θα τα παρακρατήσουμε. Εξετάζοντας το παράρτημα της έκθεσης βλέπουμε ότι ε, τα προαπαιτούμενα είναι ε, στη διακριτική ευχαίρεια του Προεδρείου. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ε, κάτι που αντίκειται στον εσωτερικό κανονισμό. Θα πρέπει να αποκατασταθεί αυτό το σφάλμα και ελπίζω ε, να μην αναγκαστώ ε, να ε, καταφερθώ με πολύ άσχημο τρόπο εναντίον αυτής της διάταξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τους μεταφραστές γιατί βοήθησαν την Google να δημιουργήσει το Google Translate και να έτσι τελικά να μεταφραστεί πανεύκολα σε 28 επίσημες γλώσσες. γλώσσες προτείνω να τους ζητήσουμε εθελοντικά να συμβάλλουν στον προϋπολογισμό του θεσμικού μας οργάνου και έτσι θα καταλάβουν ότι δεν θα πρέπει απαραίτητα να έχουν δουλειές μεσαίας τάξης με πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Σε κάθε περίπτωση τα τρέχοντα έξοδα είναι μεγάλα και διάφορα άλλα θέματα έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν σε, αυτή την, σε αυτό το εγχείρημα ε, που ενίοτε ήταν αρκετά ε, σκοτεινό και μη κατανοητό. Ελπίζω αύριο να εγκριθεί η έκθεση στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Κύριε Ζουροπή, λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Μαγκενές. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Τάραντ, τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό του 2017. Καλή είναι η θέση του και ισορροπημένη και πιστεύω ότι βοήθησε πάρα πολύ προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε έναν προπολογισμό που ήδη από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για μια επταετή περίοδο έχει περικοπεί κατά 4% και 1% ετησίως προβλέπει ε, οικονομίες από τις δαπάνες προσωπικού. Εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε όσο γίνεται πιο οικονόμοι με τα χρήματα των φορολογουμένων από το 20% που κανονικά έχουμε ε, αύξηση στις δαπάνες, στις διοικητικές. Το μειώσαμε σε 19,17% και αυτό είναι πρωτοφανές. Θυμάμαι τα τελευταία 8 χρόνια δεν είχαμε ποτέ τέτοια στοιχεία. αυξάνονται οι δαπάνες για την ασφάλεια κατά 0,6%, δηλαδή χαμηλότερα από το τιμάριθμο. Και αν δούμε και τις τακτικές δαπάνες και τις συγκρίνουμε, είναι 1,4%. Γενικά είναι πάρα πολύ φιδωλός ο προϋπολογισμός, πάρα πολύ συνετός και θα παρακαλούσα συναδέλφους ε, να ε, αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που έχουμε ο καθένας για οικονομίες. Υπάρχουν πολλοί τομείς ακόμα με ανώτατα αγορία και δεν θα πρέπει να τα εξαντλούμε κάθε φορά, ε, κάθε μέρα σε κάθε περίπτωση. Έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε ελεύθερα αποφάσεις και αυτή είναι και η ομορφιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υπάρχει μεγάλη ευθύνη που φέρει ο κάθε μεμονωμένος ευρωβουλευτής ε, πώς θα χειρίζεται τις δαπάνες του. Είτε δουλεύει πολύ είτε δουλεύει λίγο ε, είναι ελεύθερη η εντολή μας και κατά συνείδηση μπορούμε να αποφασίσουμε ο καθένας. Έχουμε μεγάλο περιθώριο. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Ντονάνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Τάραντ που πραγματικά άκουσε τους σκιώδεις ηγητές και τους αφογκράστηκε και πήγε σε σωστή κατεύθυνση η έκθεση. Εργαστήκαμε με ταχύς ρυθμούς μετά το πένθος το οποίο μας βήθησαν οι επιθέσεις στις Βρυξέλλες και καταλήξαμε στην κατάσταση προβλέψεων για το 2017 που νομίζω ότι σήμερα είναι και λογικό και ισορροπημένο. Τώρα ε, αυτό δεν συνεπέρνει τα πλήθη όταν συζητάμε ε, για τα τρέχοντα καθημερινά θέματα, αλλά στα θεσμικά όργανα αυτό έχει σημασία. Ε, θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω την ικανοποίησή μου που συγκρατήσαμε τις τρέχουσες δαπάνες αύξηση 0,14%. Θα πρέπει να απορροφηθούν και οι δαπάνες εκεί της πολυγλωσσίας. Μετά ε, την ε, ένταξη των γοεδελικών και θέματα ασφαλείας επίσης έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλω να επιμείνω στην ανάγκη να παραμείνουν χωριστές ε, οι δαπάνες που αφορούν τις επενδύσεις από τις λειτουργικές. Δεν υπάρχει αλλιώς διαφάνεια και ορατότητα στο προπολογισμό αν δεν διαχωριστούν οι δαπάνες. Υπάρχει τρέχουσα λειτουργία, οι λειτουργικές δαπάνες που είναι τα καθημερινά και οι επενδύσεις που αφορούν το μέλλον. Και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να το έχουμε υπόψη μας για τους μελλοντικού προπολογισμού. Δύο λεπτά ο κύριος Τόρβαλτς. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και το επόμενο ευχαριστώ πηγαίνει στον εισηγητή του φίλου μου τον κύριο Ταραντ. Η διαδικασία για το σχέδιο κατάστασης ε, προβλέψεων για το 2017, για τις προβλέψεις όδου και των ουσιαστικά θα πρέπει είναι διαφανές ή θα έπρεπε να είναι διαφανές. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διέπει αυτά τα θέματα διαφάνεια, τουλάχιστον αυτό λέμε συνήθως στην πατρίδα μας. Η αλήθεια είναι ότι ο προπολογισμό για το Κοινοβουλίο είναι αδιαφανής ε, ως ένα βαθμό και αυτό δεν είναι αποδεκτό και υπάρχουν πολλά διαρθρωτικά προβλήματα. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των ε, ειδήσεων και των σημερινών δαπανών. Ε, δεν ε, υπάρχουν πληροφορίες για τα έκτακτα έξοδα, ούτε για το πώς χρησιμοποιούνται οι διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που έχουν προβλεφθεί. Αυτό ήδη έχει δημοσιευτεί στο 1494. Σεμπάστια Κρίστιαν ε, Μπαράντ γεννήθηκε ε, στο Στρασβούργο γύρω το 1457. Το 1494 ε, δημοσίευσε ένα βιβλίο, το πλοίο των τρελών. Εκεί ουσιαστικά θεωρεί ότι τους τρελούς τους ε, συμπεριφέρονται με ένα διαφορετικό ε, τρόπο όμως ε, αύριο εμείς θα καταψηφίσουμε, δεν θα είμαστε μέρος ενός πληρώματος χωρίς να ξέρουμε πώς θα πρέπει να προλογείται το πλοίο σε επικίνδυνα νερά και ένας καλός λόγος ε, για αυτή την ε, προσέγγιση είναι επειδή βλέπουμε να μεγενθύνεται η έλλειψη εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να το διορθώσουμε αυτό. Θα ζητήσουμε περισσότερη διαφάνεια και θα το κάνουμε αυτό τους επόμενους μήνες για την τελική ψήφιση του προπολογισμού τον Οκτώβριο. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό για τον κύριο Ομερζά. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου και εγώ να χαιρετήσω το έργο του εισηγητή. Δεν ήταν εύκολο το έργο του. Με αυτόν τον προπολογισμό για την εκπόνησή του είχαμε μια τριπλή απέτηση. Την απέτηση να διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία, να την προστατεύσουμε, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ασφαλείας και κυρίως μια απέτηση να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά τώρα το να δώσουμε το καλό παράδειγμα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το έχουμε πάει και καλύτερα. Πιστεύω ότι κάποιες δαπάνες δεν είναι χρήσιμες και κυρίως έχω κατά νου την ε, ανακαίνιση των γραφείων ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, έχω κατά νου και ορισμένε δαπάνες που αφορούν τη μεταφορά των ευρωβουλευτών. Όμως, η ουσία είναι αλλού. Η ουσία έγκυται στη δυνατότητα να ενισχύσουμε την νομοθετική ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Και πρέπει να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω ε, ουσιαστικά αυτές τις μειώσεις που έγιναν σε σχέση με τη μετάφραση ενώ ομόφωνα στην ομάδα μας είχαμε συμφωνήσει να διατηρήσουμε αυτή την πίστοση. Και επίσης ε, θεωρώ ότι στην έκθεση αυτή θα μπορούσαμε να έχουμε και τη μετάφραση στην νοηματική. Θα ήταν θετικό κάτι τέτοιο και ελπίζω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει στο εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ μισή λεπτό για τον κύριο Φερνάντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη θετική δουλειά που έκανε, για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε Συγχαρητήρια σας αξίζουν και γι' αυτό υπερψηφίζουμε την έκθεση. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως ε, μιλάμε για το 94% για τις επενδύσεις και μόνο 6% για όλα τα διοικητικά έξοδα. Και κατόπιν ε, μιλάμε και για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου είναι σαν να μιλάμε για το 1 πέμπτο αυτών των διοικητικών δαπανών και πρέπει να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να έχουμε μια κατάλληλη νομοθεσία υψηλής ποιότητας ποιότητας και γι' αυτό χρειαζόμαστε το ελάχιστο αλλά να επαρκεί δηλαδή τα τεχνικά μέσα και τους ανθρώπινους πόρους. Πέραν αυτού όλοι περασπίζουμε την πολυγλωσία, την πολυμορφία και βέβαια την ασφάλεια, την ασφάλεια όσων εργάζονται εδώ. Επίσης θέλουμε και συστήματα που να μας διασφαλίζουν εναντί των κυβερνοεπιθέσεων και χρειαζόμαστε όλα τα απαραίτητα μέσα να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Εμείς θέλουμε αυστηρό προπολογισμό και εργαζόμαστε γι' αυτό έναν υπολογισμό επαρκή που να μας δίνει τα απαραίτητα μέσα για να απαντήσουμε θετικά στις προκλήσεις που έχουμε ενωπιών μας. Τις προκλήσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτή την έκθεση. Δεν είναι ιδανική, αλλά είναι εφικτή και ουσιαστικά συμβάλλει στο να βελτιώνει την αρχική πρόταση που μας δόθηκε από το Γενικό Γραμματέα. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για ένα μισή λεπτό. Κύριος Βιώτη. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποιες πτυχές αυτού του προπλογισμού. Ευχαριστώ κυρίως τον εισηγητή και όσους συνεργάστηκαν μαζί του. Εγώ πιστεύω ότι η δουλειά που κάναμε στην Επιτροπή με όλες τις ομάδες μας επέτρεπε να έχουμε πολύ περισσότερες εξοικονομήσεις. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια ευρύτερη δουλειά. Νομίζω ότι οι νέε δαπάνε για την ασφάλεια και είμαστε πεπισμένοι όχι τόσο για την μας ασφάλεια, για την ασφάλεια των συνεργατών μας. Είναι απαραίτητες δαπάνες ε, βεβαίως, αλλά είναι κάπως υπερβολικές. Εγώ νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να θέσουμε τέλος το θέμα της ασφαλείας για να ε, δικαιολογούμε οποιοδήποτε είδος δαπάνης. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που θα αναφέρω ε, με τους οδηγούς. Νομίζω ότι γίνεται ένα πολύ μεγάλο λάθος αξιολόγησης και ένα λάθος στον υπολογισμό. Πρέπει να δώσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες γιατί και ο προπολογισμό έχει να κάνει με το τι απαιτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, ότι θέλουν έναν πιο εξισορροπημένο προπολογισμό που θα εξοικονομεί περισσότερα χρήματα. Ο κύριος Μπενίτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να καταγγείλω την έλλειψη σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίστηκε το θέμα αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν φταίει βέβαια ο συγητής το Κοινοβούλιο το μόνο που κάνει είναι να ακολουθεί τις προσταγές στην Επιτροπή και είχε μία μέρα μόνο να αξιολογήσει, ε, στη διάθεσή του να αξιολογήσει τις εκθέσεις. Με την κρίση που διασχίζει, που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη λιτότητα που απαιτείται τα κράτη-μέλη θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει υποδειγματική συμπεριφορά και τα θεσμικά όργανα έπρεπε να δίνουν το καλό Παράδειγμα, δεν υπάρχει ορισμός του έκτακτου εξόδου. Πληρώνονται εισιτήρια αεροπορικά σε θέση business ε, και διάφορες άλλες πατάλες και εξόφθαλμες ε, υπερβάσεις θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Ζητούμε να υπάρχει μία μόνο έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το να υπάρχουν διάφορες έδρες ε, και τόσες πολλές μετακινήσεις ε, σημαίνει τεράστια έξοδα. 180 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στοιχίζει αυτό το πηγενέλα. Και θα ήθελα να προτείνω την έδρα να την έχουμε στη, ε, στην πατρίδα μου, στον Μπιλμπάο. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Φέντεχοφσκι για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία να, για να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδους εισηγητές για την πολύ καλή του συνεργασία και θέλω να εκφράσω μια πρωτότυπη ιδέα που δεν έχει υποθεί σήμερα εδώ. Ίσως δεν το έχετε καταλάβει και δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία και ως εκ τούτου υφίσταται και μεγαλύτερες απειλές. Επομένως, θα πρέπει στο μέλλον όχι μόνο να διασφαλίσουμε ότι έχουμε επαρκή προπολογισμό για θέματα ασφαλείας, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ευέλικτοι, να είμαστε σε θέση να υιοθετήσουμε μέτρα ad hoc, επιτόπου, τα οποία αποδείχτηκαν απαραίτητα φέτος. Και ε, θέλω να το τονίσω αυτό. Δεν έχει κανένα νόημα να συζητούμε πόσο αποτελεσματικό είναι να εξοδεύουμε τόσα χρήματα για να πηγαίνουμε και να επιστρέφουμε από και προς το Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες. Σε πάση περιπτώσει αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν έχουμε ούτε καν δύο κτίρια, έχουμε τρία κτίρια. Αλλά όσο και να έχουμε πρέπει να έχουμε παρκή ασφάλεια, να το διασφαλίσουμε αυτό. Έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορούν να δουλέψουν σε συνθήκες ασφαλείας. Τώρα, αν συζητούμε για το ποια εξοικονόμηση θα κάνουμε, κάνουμε ε, καταργώντας μία από τις έδρες, ε, τότε δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτό. Γιατί θα πρέπει να συζητούμε για ισολογισμούς, για ισορροπημένο προϋπολογισμό, λυσμένο. Το θέμα είναι πώς ξοδεύονται τα χρήματα και θα πρέπει να τα αξιοποιούμε τον καλύτερο δυνατό ε, τρόπο. Ευχαριστώ κύριο Μάνκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε, όταν ε, συντάσσει κανείς ένα σχέδιο προϋπολογισμού, το πιο απλό είναι να πολλαπλασιάσει το περσινό υπολογισμό με το συντελεστή του πληθωρισμού ή, με κάτι τέτοιο. Και αν το επαναλαμβάνει κανείς αυτό κάθε χρόνο, τελικά θα καταλήξει σε, μη, σε ανακρίβειες και σε αναποτελεσματική χρήση πόρων. Ο πληθωρισμός πρόσφατα ήταν πολύ χαμηλότερος από τον προϋπολογισμό που είχε ε, ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του αρχικού σχεδίου και αυτό, αυτές οι διορθώσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουμε να βελτιώσουμε την παρέμβασή μας και ελπίζουμε μετά την αυριανή ψηφοφορία να καταρτίζονται όλοι οι προϋπολογισμοί για όλες τις χρήσεις της οικονομικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο σε συμφωνία ε, με ε, τα δέοντα και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τους πόρους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ κύριος Ντόρφμαν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τους και εισηγητές ειλικρινά γιατί νομίζω ότι είναι γερό το αποτέλεσμα και που μπορούμε και προς τα έξω να το υπερασπιστούμε. Στον προπολογισμό ενός θεσμικού οργάνου σαν το δικό μας θα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Από τη μια οι πολίτες απαιτούν να είμαστε συνετοί και φρόνιμοι στη χρήση μας και να προσπαθούμε ε, να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά ε, με όσο γίνεται λιγότερες δαπάνες. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα ε, στα ταξίδια και τις αντιπροσωπείες που έχουμε να σκεφτούμε πόσοι ε, θα πηγαίνουν, πόσες γλώσσες χρειαζόμαστε και αντίστοιχα να κάνουμε και οικονομίες και συμφωνώ με αυτό. Από την άλλη όμως υπάρχει και το θέμα της ποιότητας της κοινοβουλευτικής δουλειάς που θα πρέπει να είναι δεδομένη και εξασφαλισμένη και αυτό έχει να κάνει και με τους υπαλλήλους που χρηματοδοτούμε με τα πολιτικά κόμματα ευτυχώς καταφέραμε και στον προπολογισμό ε, της κοινοβουλευτικής ε, Ένωσης που ε, είμαι πρόεδρος να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότησή της γιατί είναι σημαντικό για τη δημοκρατία και για τη δημοκρατική συζήτηση. Καλό είναι λοιπόν να κάνουμε μια χρηστή διαχείριση. Συμφωνώ με τον προπολογισμό που προτείνεται και ελπίζω και εύχομαι αύριο να τον υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. And thank you. We now move to catch... Ευχαριστώ. Πάμε στη διαδικασία Κασιάη. Ο κύριος Νεκρέσκου πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση για την κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2017 είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση. Υπάρχουν κάποια κονδύλια που χρειάζεται το Κοινοβούλιο για να λειτουργεί και σημαντικά μέτρα ε, προτείνονται για τη ε, μεγαλύτερη διαφάνεια και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της λειτουργίας μας. Η δημοσίευση του προπολογισμού στην ιστοσελίδα είναι μια κίνηση καλή θέληση για να δείξουμε ότι θέλουμε να τα βλέπουν όλοι οι πολίτες. Μια ισχυρή δημοκρατία προποθέτει ισχυρό κοινοβούλιο. Ένα κοινοβούλιο που να επικοινωνεί με τους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμο, όχι μόνο στι Βρυξέλλε ή στο Στρασβούργο, παντού στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό λοιπόν δεν πιστεύω ότι είναι καλό να επιβάλλουμε και νέες διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Για την Ανατολική Ευρώπη ήδη υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί και αυτό δεν είναι καλό. Και μιλώ για τους εργαζομένους που παίρνουν περισσότερα, λιγότερα χρήματα. Ο κύριος Μαριάς παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στα πλαίσια των προβλέψεων για τα έσοδα και τις δαπάνες του Κοινοβουλίου για το 2017 η ασφάλεια και η κυβερνοασφάλεια έχουν οριστεί ως οι πρωταρχικοί στόχοι για τον προϋπολογισμό. συγκεκριμένα υπάρχει πρόβλεψη για συνολική αύξηση του προϋπολογισμού του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου το 2017 κατά 3,9% σε σχέση με αυτόν του 2016. ενώ για την ενίσχυση της ασφάλειας απαιτούνται επενδύσεις ύψους 36,8 εκατομμυρίων ευρώ. γενικότερα οποιοδήποτε μέτρο στον τομέα της ασφάλειας θα πρέπει να προκύπτει έπειτα από αξιολόγηση των αναγκών του κοινοβουλίου και των ενδεχόμενων κινδύνων. θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει έλεγχος και στα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας καθώς και στις δημοσιονομικές επιπτώσεις που θα έχουν. τέλος θα πρέπει να παρουσιάζεται με ακρίβεια η εξέλιξη του προϋπολογισμού του κοινοβουλίου για κάθε έτος προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται. διαφάνεια λοιπόν σε όλα και για όλα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Νιριάντα, ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να αναφερθώ στην προτεραιότητα για τα Ιρλανδικά και για το γεγονός ότι δίνεται υποστήριξη στην Ιρλανδική γλώσσα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η γλώσσα μας, πρέπει να την προωθήσουμε και θα πρέπει να μπει στο ίδιο επίπεδο με όλες τις άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν μπορέσαμε να στείλουμε ένα μήνυμα για το πόσο σημαντική είναι η ταυτότητά μας και πώς αναγνωρίζεται εδώ σε αυτό τον οίκο. Θα ήθελα να καλωσορίσω και το γεγονός ότι τα 3,7 εκατομμύρια έχουν τεθεί για το σκοπό αυτό, για να ξεκινήσουμε και τη διαδικασία πρόσληψης έτσι ώστε να μπορούσαμε να παράσχουμε γλωσσικές υπηρεσίες. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα, μπορούσαμε να, θα να υποφεληθούμε από τις γλωσσικές υπηρεσίες στην Ιρλανδική, γιατί έχω δώσει αγώνα για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριος Βίγκας. Εμείς σε αυτή την έκθεση βλέπουμε ότι είναι σημαντικό να διατηρούμε την ισορροπία, όμως ε, θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε αποκλεισμό. Εμείς ε, όμως δεν συμφωνούμε με την λιτότητα. Μιλούμε πάντοτε για μείωση των πόρων και πάντοτε στους ίδιους τομείς. Είμαστε ευαίσθητοι στο θέμα της ασφάλειας, αλλά δεν θεωρούμε ότι πρέπει να υπερβάλλουμε και κάθε φορά αυτό το κοινοβούλιο μοιάζει με φρούριο ή με φυλακή. Δεν καταλαβαίνουμε και τη μείωση του προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα θέλουμε να δίνουμε όλο και μεγαλύτερη σημασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης ε, δεν συμφωνούμε σε αυτά που λέγονται ε, για τις υπηρεσίες μεταφορών ε, και θα πρέπει ουσιαστικά το Κοινοβούλιο να προωθεί τα δικαιώματα των εργαζομένων του. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ακούσουμε τον εισηγητή, τον κύριο Τάραντ, για να κλείσει αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ενδιαφέρουσα όσο και ουσιαστική η συζήτηση και τα σχόλια και οι ομιλίες που ακούσαμε. Καλή εντύπωση έκαναν στον ίδιο το συνεχίτη τον υποφαινόμενο. Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια, είμαστε καμιά εικοσαριά βουλευτές και ακούμε πολιτικές απόψεις και γνώμες που θα καθορίσουν την αυριανή ψηφοφορία. Και όπως σας είπα, εγώ θα δεχτώ το δημοκρατικό αποτέλεσμα. Είμαι έτοιμος και για τις ε, διαπραγματεύσεις τελευταίας στιγμής, αν θέλετε τώρα ε, νυχτιάτικα να προσπαθήσουμε κάτι να βελτιώσουμε. Η έκθεσή μου επιζητεί ε, συμβιβασμό μεταξύ διαφόρων θεσμικών οργάνων, ε, ε, πολιτικών ομάδων και προσωπικότητων. Και είχα τη χαρά και την ευτυχία να γνωρίσω διάφορες τέτοιες ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Καμία έκθεση τέτοιου είδους δεν μπορεί να είναι ιδανική. Χωράει πολλές επικρίσεις και γελιοποιήσεις και αμφισβητήσεις. Αυτή τη στιγμή όμως αυτή την έκθεση διαθέτουμε και αύριο πρέπει να την ψηφίσουμε. Τι να κάνουμε, ας την ψηφίσουμε και είδομεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή για τον προϋπολογισμό.